Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Καλό σας απόγευμα. ξεκινήσουμε διότι έχουμε φορτωμένη διάταξη εδώ. Γιατί αρκετοί από τους ε, παρεμβαίνοντες ε, θα μιλήσουν μέσω βίντεο link, το οποίο δεν είναι τεχνικός εύκολο. Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Θα κάνω μία πολύ σύντομη εισαγωγή και βεβαίω με κάθε σεβασμό προς τις αρχές της Βενεζουέλας γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας ε, εξετάζει με μεγάλο ενδιαφέρον και ανησυχία την κατάσταση στην Βενεζουέλα. Θα ήθελα να βεβαιώσω τις αρχές της Βενεζουέλας προς αρχές προς οποίες με συγχωρείτε απευθύναμε πρόσκληση και δεν ανταποκρίθηκαν ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση παρέμβαση στα εσωτερικά θέματα της Βενεζουέλας. Θα ήταν πολύ καλό και όμορφο η κάθε χώρα να προχωρεί στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας, όμως η Βενεζουέλα δεν μπορεί να μείνει εκτός της επιτήρησης που πραγματοποιεί η Επιτροπή μας για τα ανθρωπίνα δικαιώματα γιατί εξετάζουμε περιπτώσεις οι οποίες, ε, οι οποίες είναι πιθανές παραβιάσεις τέτοιων ανθρωπίων δικαιωμάτων. Αυτή είναι η άποψή μου. Διότι όταν έχουμε πολιτικούς ηγέτες της αντιπολίτευσης στη φυλακή, είναι πολύ κακό σημάδι όπως γνωρίζουμε. Και σε σχέση με τα εκλογικά αποτελέσματα, τους πολίτες και τους θεσμούς, αυτό που είναι κανονικό σε μια δημοκρατία επί της αρχής θεωρητικός είναι το σύστημα που έχει οθετήσει η Βενεζουέλα. Το κανονικό λοιπόν είναι όλες αυτές οι αρχές της αντιπολίτευσης για παράδειγμα να προστατεύονται από τον νόμο. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι μόνο να διοργανώνουμε την εκλογική αναμέτρηση αλλά πρέπει να σεβόμαστε τις δημοκρατικές αρχές σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να εγγυάται η συμμετοχή των οργανισμών και των φορέων και των πολιτικών κομμάτων στη διαδικασία. Και δεν μπορεί το κράτος ε, να ενοχοποιεί και να αποδίδει εγκληματικές ε, πράξεις ή κατηγορίες ή προθέσεις κατά των ε, ηγετών της αντιπολίτευσης. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πεπισμένοι όπως και μεγάλο μέρος της κοινωνίας Βενεζουέλας ότι αυτή η ακραία προσέγγιση που έχει επιλέξει η Βενεζουέλα δεν είναι η καλύτερη λύση. Και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να συμμετάσχω σε κάποιο είδους conspiracy theory κατά της ε, Βενεζουέλα. Εγώ το λέω ως φίλη και σύμμαχος της χώρας αυτής. Δεν θέλουμε να δώσουμε μαθήματα, ούτε να παραδειγματίσουμε. Αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς ε, της χώρας να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ενός, ε, μιας δημοκρατικής χώρας, ε, ενός κράτους δικαίου. Και πιστεύω εκπροσωπώντας την μεγάλη πλειοψηφία της αίθουσα. Νομίζω ότι πρέπει να απελευθερωθεί ο Δήμαρχος του Καράκας και των υπολείπων εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων αντιπολίτευση. Και έτσι έπραξε ως σύσταση και τον περασμένο Αύγουστο η συγκεκριμένη Επιτροπή των ε, Ηνωμένων Εθνών Λεπόλτο Λόπεθ και ε, κύριος Θεβάγιος είχαν αναφερθεί ρητά είχε ζητηθεί από την ε, κυβέρνηση της Βενιζουέλα να σε απελευθερώσει και η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών με μεγάλη στα θέματα της Νοτιοαμερικής είπε ότι αυτό δεν είναι συμβατό με τα διεθνή ε, με, με το διεθνές κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλούμε για προληπτικές ε, κρατήσεις ε, με δίθεν ποινικέ κατηγορίες το οποίο στην ουσία προκαταλαμβάνει την οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου. Χρειαζόμαστε λοιπόν αναλογικότητα και μια λογική προσέγγιση θα έλεγα και συνετή προσέγγιση. Θα μας ε, άρεσε, θα θέλαμε να εγκατασταθεί μια πραγματική πολιτική διαβούλευση συζήτηση στη Βενεζουέλα και αλλά αυτό να αναπτυχθεί με σεβασμό προς κάθε δυνατή επιλογή. Δεν θέλουμε να υπάρξουν θύματα, αθώα θύματα μιας ε, κλιμάκωσης και απέναντι στο αίτημα αυτό να απελευθερωθούν οι πολιτικοί αυτοί κρατούμενοι της Βενεζουέλα, ίσως αυτό να μην τον ενδιαφέρει τον πρόεδρο Μαδούρο, εμάς όμως μας ενδιαφέρει και θα επιμείνουμε. Και στον ερχόμενο μήνα εγώ θα συμμετάσχω σε αποστολή του Ερωικού Κοινοβουλίου και θα διαβιβάσω το αίτημα αυτό προσωπικά στις αρχές Βενεζουέλας. Δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό πρόγραμμα προσωπικά του Πρόεδρου, αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα να υπερασπιζόμαστε τα θύματα, τους κρατουμένους αυτής της άδικης μεταχείρισης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δύο ψηφίσματα έχει ήδη εκφράσει όλα τα όσα σας λέω και είναι απολύτως απαραίτητο, απαραίτητο αντικειμενικά να εξετάσουμε ποια είναι η κατάσταση, η πραγματική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε λοιπόν καλεσμένου σήμερα πολύ σημαντικού οι οποίοι θα μα δώσουν μια πλήρη εικόνα και αντικειμενική, ο καθένα από τη δική του οπτική γωνία, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα. Έχουμε λοιπόν διάφορους ε, συνεισφέροντε, κάποιους ζωντανά, κάποιου μέσω βίντεο διάσκεψης, θα μπορέσουμε αν θα, θα εξετάσουμε αν θα μπορέσουμε να, να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο μας με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο ώστε να έχουμε και παρεμβάσει από την αίθουσα αλλά καθότι περιμένουν κάποιοι ήδη για τα βίντεο link θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Ντέλσα Σολορθάνο μέλος του Κοινοβουλίου της Λατινικής Αμερικής η ε, κυρία Σολορθάνο παρακαλώ έχει το λόγο Δεν tratando de hacer la conexión. Δεν ξέρω ποιος προσπαθεί να κάνει τη σύνδεση, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ας συνεχίσουμε και στο μεταξύ θα, λόγω το, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ασίφ που πρέπει να φύγει και νωρίτερα. Bueno, pues mientras siguen intentando conectar. Περιμένοντας την ε, σύνδεση με την κυρία Σολορθάνο θα δώσω το λόγο στον κύριο Καμπρέρα, ο οποίος ε, εκπροσωπεί τα θύματα της ε, Γκουαρίμπα και του Γκόλπε Κοντινουάδο. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ονομάζομαι Καμπρέρα Είμαι ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής των Θυμάτων της Γκουαρίμπα και του Γκόλπε Κοντινουάδο. Πρόκειται για μη κυβερνητική η οποία περιλαμβάνει ε, όλα τα θύματα που ε, πλήγησαν το 13 και το 14. Ο κύριος Λουίς Ντουράν και ο κύριος Καρέρο είναι μέλη της Επιτροπής μαζί μου. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να είμαι εδώ στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να σας πω τι ακριβώς συνέβη στη χώρα μου τα τελευταία χρόνια και να αποδοθεί δικαιοσύνη στις οικογένειες και στα θύματα. Εγώ δεν είμαι πολιτικός ηγέτης, ούτε εκπροσωπώ πολιτικές οργανώσεις. Είμαι μία η μητέρα που έχει μία κόρη 19 μηνών που είδε πώς πλήττονται τα θύματα σε επίπεδο μικρών παιδιών μέχρι τριών ετών. Εμείς που συμμετέχουμε σε αυτή την Επιτροπή ε, είμαστε θύματα δύο φορές. Καταρχήν γιατί πολλοί έχασαν ε, τα κοντινά τους πρόσωπα από την πολιτική βία. Για παράδειγμα ο Λουίς Ντουράν που βρίσκεται στην αίθουσα είναι ένα από τα θύματα που σκότωσαν το παιδί του, το καρατόμησαν όταν προσπάθησε να παρέμβει και όταν περνούσαν μοτοσυκλετιστές που συμμετείχαν σε μια διαδήλωση. Ο κύριος Όσκαρ Καρέρο επίσης ήταν ε, θύμα ε, ακριβώς επειδή σε ένα κρατήδιο ε, έσκασε μία βόμβα σε ε, ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε φαρμακευτικά σκεύη. Σκευάσματα, με συγχωρείτε. Δεύτερον, Υπήρξαμε θύματα γιατί έγινε πολιτική χρήση αυτών των γεγονότων από διεθνείς οργανώσεις και ΜΜΕ στις δικές μας περιπτώσεις. Κύριοι βουλευτές, όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέτε ότι τα 43 θύματα το 14 ήταν φοιτητές και ε, συμμετέχονται σε ειρηνικές διαδηλώσεις κατά του Νικολάς Μαδούρο, εμείς νιώθουμε μεγάλο θυμό, όχι μόνο γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο ψέμα και χειραγώγηση, γιατί θεωρούμε ότι χρησιμοποιήθηκε ο πόνος μας για να προσπαθήσουν μερικοί να καρποθούν πολιτικά την κατάσταση. Η αλήθεια, κύριοι βουλευτές, είναι ότι 35 από τα 43 άτομα που έχασαν τη ζωή τους είναι πρόσωπα που συμμετέχουν σε δύο εκδηλώσεις στις 12 Φεβρουαρίου το 2014 έβαλαν πραγματικά θανάσιμες παγίδες στις δημόσιες οδούς και προσπάθησαν να στήσουν χαρακόμματα και να πυροβολήσουν. Ε, έκαψαν κέντρα υγείας και δημόσια ιδρύματα και όλα αυτά για να προσπαθήσουν να αναγκάσουν την εθνική κυβέρνηση να αντιδράσει είχαμε 878 τραυματίες και χιλιάδες ανθρώπους που είδαν να πλήττονται τα δικαιώματά τους ως προς την υγεία, την εκπαίδευση, την ελεύθερη κυκλοφορία και την ελεύθερη ε, διακίνηση. Όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλα φόρα μιλάμε για την απελευθέρωση των ε, κρατουμένων, μέσα στα πλαίσια αυτών των βίαιων εκδηλώσεων και μιλάμε για πολιτικούς κρατούμενους, στην ουσία ε, προωθούμε την ατιμορρησία για ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για βίαιες εκδηλώσεις και καταπατώνται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει το κοινοβούλιο σας να γνωρίζει ότι πέρα από τον ε, Λεοπόλτο Λόπες και τον ε, κύριο Σεμπάγιος Υπάρχει και ο Έλβις Τουράν, ο οποίος ήταν ε, θύμα δύο εκδηλώσεων, έχασε τη ζωή του και άφησε ένα μικρό παιδί. Ο κύριος Γκονσάλες, ε, ο ε, εισαγγελέας, ο δημόσιος κατήγορος, επίσης έχασε τη ζωή του. Προσπαθούμε να ε, δούμε τι ακριβώς συνέβη σε ένα από αυτά τα ε, χαρακόμματα όπου έχασε τη ζωή του και ένας άλλος άνθρωπος που άφησε τέσσερα ορφανά. Ο Χωσέ Κολίνας, ο οποίος άφησε στη ζωή τη γυναίκα του η οποία ήταν έγκυος. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε και ένα άλλο θύμα το οποίο χάσε τη ζωή του αφού πυροβολήθηκε στο κεφάλι και άφησε μία οικογένεια ορφανή. Όλα αυτά έγιναν πέρσι στη Βενεζουέλα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τα πραγματικά θύματα. Ελπίζω τα ονόματά τους να αναφέρονται στα, στις συζητήσεις του Κοινοβουλίου και ελπίζω να τιμήσετε τα θύματα της Γκουαρίμπα και να εισακουστούν οι εκκλήσεις μας σε αυτή την ακρόαση. Εξ ονόματος της Επιτροπής μας θα θέλαμε να μην χρησιμοποιηθεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μέσο χειραγώγησης. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις και διαδηλώσεις ειρηνικού χαρακτήρα, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη βία και τα εγκλήματα υπέρ των ειρηνικών δίθεν εκδηλώσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ε, πραγματικές προθέσεις των πολιτικών κομμάτων όταν οργάνωσαν τις ε, βίες αυτές διαδηλώσεις από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2014. Οι πραγματικές προθέσεις που γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς ε, με βάση τα, αυτά που είπε ο κύριος Λόπες, όταν τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος πότε θα τελειώσουν όλα αυτά και απάντησε ο κύριος Λόπες, γνωστός δημοσιογράφος, όταν βγάλουμε από την εξουσία όλους αυτούς που βρίσκονται εκεί. Δεν θα πρέπει να κολλησιεργούμε όπως έκαναν ορισμένοι πολιτικοί, πολιτικοί ηγέτες και ΜΜΕ, καθώς και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα θέλαμε να ε, θεωρηθούν αυτοί οι θήτες ότι πραγματικά υπήρξαν θήτες οι οποίοι έπληξαν την κοινωνία μας και θα πρέπει να τιμωρηθούν. Επίσης, με τη δράση μας αυτή θα θέλαμε να μην υπάρχει ατιμορρησία και να υπάρξουν να υπάρξει πραγματική τιμωρία για τους θύτες. Επίσης, να υπάρχει σεβασμός και αλληλεγγύη προς όλα τα θύματα, γιατί χάσαμε αγαπημένα πρόσωπα. Δεν μπορούν αυτοί που χρησιμοποιούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, για να χειραγωγήσουν πολιτικές πράξεις, να ε, περάσουν ατιμωρητοί στην ιστορία. Έχουμε Σα ευχαριστώ, σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Έχουμε ήδη συνδεδεμένη την κυρία Ντέλσα Σολορθάνο που είναι εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου τη Λατινική Αμερική. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κυρία Ντέλσα Σολορθάνο. Ίσως θα μπορούσαμε να χαμηλώσουμε λίγο και τα φώτα, λέει η Πρόεδρος, για να βλέπουμε καλύτερα την οθόνη. Όποτε θέλετε, ξεκινάτε. Είμαι η Ντέλσα Σολόρσανο, είμαι μέρος de la Unidad Democrática coordinar la política de derechos humanos. A lo largo de todos estos un momento, un momento, un momento. Ένα λεπτό διακόπτει η πρόεδρος διότι έχουμε πρόεδρο με τον ήχο. Οι διερμηνείς δεν μπορούν, δεν μπορούν να διερμηνεύσουν υπό τις συνθήκες αυτές λέει η πρόεδρος και έχει δίκαιο. Φοράτε το μικρόφωνο σας ή το έχετε μπροστά σας αν μπορείτε να πλησιάσετε λίγο εμείς οι Ισπανόφωνοι καταλαβαίνουμε καλά λέει ο Πρόεδρος αλλά οι υπόλοιποι για να μπορέσει να διερμηνευτεί η παρέμβασή σας Δεκαοχτώ χρόνια ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Έχουμε πολύ κακό ήχο από τη διερμηνία. Πολύ κακό ήχο de la Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο δυστυχώ. Ούτε καν στα ισπανικά λέει η πρόεδρο. Δεν μπορώ εγώ να σα παρακολουθήσω καλά. Έχουμε συνεχεί διακοπέ. Δεν ξέρω αν έχετε τεχνικό εκεί μαζί σα. Να του διαβιβάσετε παρακαλώ ότι έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Ειδικά για όσους δεν σας παρακολουθούν απευθεία στα ισπανικά είναι αδύνατον. Εντρεκόρτ. Έχουμε διακοπές συνεχής. Bueno, el Parlamento Europeo tiene mucho que mejorar en términos το κοινοβούλιο είναι αλήθεια ότι λέει η Πρόεδρος ότι πρέπει πολύ να βελτιώσει την κατάσταση τεχνικός φως. Μας συμβαίνει συνεχώς, όχι μόνο με τις συνδέσεις ε, της live με τη Βενεζουέλα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Αβελίδο που είναι υπεύθυνο ε, για τα εξωτερικά θέματα της Μέσα Δημοκράτικα, όποτε θέλετε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Μάρτιο το Κοινοβούλιο εξέδωσε το τελευταίο ψήφισμα του επί της Βενεζουέλα μετά τις 27 Φεβρουαρίου και τις 18 Δεκεμβρίου για να μιλήσω μόνο για τα πιο πρόσφατα. Το Κοινοβούλιο λοιπόν επί τη βάση των γεγονότων στη χώρα μας με τις επιπτώσεις που είχαμε από την κράτηση του Δημάρχου του Καράκας που αυτή τη στιγμή είναι κρατούμενος κατοίκων η ακρόαση διακόπη για τρίτη φορά την περασμένη Δευτέρα 9 Ιουνίου και από το Μάρτιο μέχρι εδώ έτσι όπως συμβαίνει και με την οικονομική και κοινωνική και πολιτική κατάσταση το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα με συγχωρείτε, έγινε πιο δυσχερές. Και το παρακολουθεί αυτό μια διαμερικανική επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την υποπτία των διεθνών οργανισμών και φορέων για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα υπό την CIDH το, η οποία παρακολουθεί το Διεθνές Εφαρμοστείο Δίκαιο. Και μιλούμε για την ασφάλεια των πολιτών, την ασφάλεια στην ουσία της λειτουργίας δημοκρατίας. Μέχρι το Μάιο του 2015 έχαναν τη ζωή τους 250 ε, και άνω χιλιάδες ε, πολίτες. Η ατιμορρησία η καμία, ο, ο, ο μηδενικός σεβασμός για τα δικαιώματα των πολιτών ή για τις, μάλλον ο πλευρά των αστυνομικών και στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών αρχών της Βενεζουέλας οδηγούν στη δημιουργία πολιτοφυλακών με παραστρατιωτικές αρμοδιότητες οι οποίες πλήττουν τα δικαιώματα των πολιτών και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Στην ετήσια έκθεση μιλούμε για 137% αύξηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταγράφονται συγκεκριμένες περιπτώσεις, 185 μάλιστα, είχαμε τον, από το κρατήδιο Μιράντα τον ε, εκπρόσωπο των ε, ε, προεδρικών εκλογών της Δημοκρατικής Ένωσης και πειραματισμού σχετικά με, τις παρα... τη δράση των παραστρατικών και παρααστυνομικών παραστυνομικών θα έλεγα αυτών οργανώσεων προκειμένου να επιτύχουν θεωρητικούς στόχους σχεδίων και παραθέτω τον καράγο, τον ε, κυβερνήτη, ότι το, πιο σημαντικό είναι να έχουμε ένα κράτος που να αποφεύγουμε ότι ο κυβερνήτης Μιράντα, δηλαδή να, να καταφέρουμε να μην διοικείται από έναν ε, ε, τόσο αντιδραστικό στοιχείο όπως το κυβερνήτη Μιράντα. Επομένως πλήττεται ο, ο κυβερνήτης ε, Μιράντα για τις αντί επαναστατικές του εντός εγωνικών αυτές θέσεις. Τον Απρίλιο ο υποψήφιος της, ε, στον πρώτο γύρο των ε, εκλογών για το Καράκα Σαβέριο Βίβας ταυτοποιήθηκε από την κυβέρνηση του αρνήθηκαν το σχηματισμό κομμάτων υπό την Μαρία Κολίνα Ματσάδο και από, την, από περασμένο έτος αυτά γίνονται με μοναδική απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου χωρίς καμία άλλη διαδικασία και συζήτηση. Αποφασίστηκε παράνομα τα μέλη του Κοινοβουλίου να μην ψηφίζονται με λαϊκή ψήφο όπως προβλέπει η νομοθεσία και γίνεται από το 1928 αλλά να ορίζονται από την αίθουσα, από το Κοινοβούλιο. Ακόμα φέτο δεν έχει δημοσιευτεί τίποτα περαιτέρω για τα μέλη του Κοινοβουλίου που θα πρέπει να του δοθεί εντολή από τι 5 Ιανουαρίου του 2016. Ο Λεοπόλτο Λόπεθ και ο Ντανιέλ Θεβάγιο αλλά και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι έχουν ήδη διακηρύξει ότι είναι σε, σε απεργία πείνα. Όλα αυτά τα μέσα ε, τα χρησιμοποιούν τακτικά και δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στην ελευθερία έκφρασης το Μάιο μετά τη δημοσίευση πληροφοριών από τον ξένο τύπο σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος της αίθουσα ε, ε, βαρύ, βαρύνεται με, ε, με συγκεκριμένα ποινικά δικήματα, αυτά δημοσιεύτηκαν σε ξένες εφημερίδες και είχαμε και την ιστοσελίδα lapatilla.com που δημοσίευσε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα ποινικά αυτά αδικήματα όμως δεν επιτράπει στη δικαιοσύνη να λειτουργήσει αυτόνομα διότι υπάρχει ε, ε, κυβερνητικό μονοπόλιο για, τις, ε, για τον τύπο, για τις εφημερίδες, και τα περιόδικα, για τα περιοδικά Επίσης ε, έχει απολέσει το σύνολο της κοινωνίας ε, την αγοραστική του δύναμη. Έχουμε τρομακτικό πληθωρισμό. Ε, έχουμε συνεχή επιδίνωση των υπηρεσιών των κρατικών και των δημόσιων. Έχουμε αύξηση της στόχιας. Έχουμε συνεχή αύξηση 3.200% και άνω των βασικών προϊόντων διατροφής Μάλιστα, εξ αυτού και η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ε, τοποθετήθηκε ότι για την σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων δεν έχει πετύχει κανένα από τους στόχους της η Κυβερνητική Επιτροπή. Επομένως, η σοβαρότητα της κατάστασης ε, στη Βενεζουέλα έχει αποτυπωθεί και από τις συνδικαλιστικές ενώσεις όπως και από τις ενώσεις εργοδοτών για τις συμβάσεις 87, 26 για τον ελάχιστο μισθό, 144 ε, για, τις, για τις τριμερείς ε, διαβουλεύσεις. Εξ ονόματος ε, του λαού της Βενεζουέλας σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την έκφραση του ενδιαφέροντος και τη στήριξη αυτής. Ας δούμε λοιπόν κατά πόσο μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την κυρία Σολορθάνο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Είμαι αντιπρόεδρος της, ε, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και συντονίζω τα ανθρώπινα, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη χώρα μας υπάρχει μεγάλη κρίση σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχουν, με συγχωρείτε, είναι κάκιστη ποιότητα ήχου, δεν μπορούμε να κάνουμε διερμηνία. No ε, να φρανσέσι. Δυστυχώς δεν σας ακούμε, λέει η ε, πρόεδρος. Ε, δεν ακούγεται καλά για τους ε, διερμηνείς. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει διερμηνία. Είναι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 ε, κόμματα με διαφορετική ιδεολογική βάση. Προσπαθούμε λοιπόν να ανταποκριθούμε με βάση τα δημοκρατικά δεδομένα στις 12 Φεβρουαρίου 2014 είδαμε ότι ε, εκρατούντο 3.167 πολίτες ε, για πολιτικούς λόγους. Μόνο οι 709 ε, πόρεσαν να απελευθερωθούν. 2.383 ε, στην ουσία κρατούνται ή εν πάση περιπτώσει στερούνται των ελευθεριών τους. 14 ε, βρίσκονται υπό ε, κατοίκο περιορισμό και 61 στερούνται της ελευθερίας τους. Και από το 2012 11 πολίτες ε, κρατούνται. Έχουμε λοιπόν αυτό τον αριθμό των πολιτικών κρατουμένων. Υπάρχουν πολιτικές διώξεις και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μανουέλ Ροσάλες ε, είναι εξόριστος. Ήταν προε... υποψήφιος για την Προεδρία το 2006, αλλά δυστυχώς στη συνέχεια η εκτελεστική εξουσία τον ε, καταδίκασε στην εξουσία και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 Siento Με συγχωρείτε γιατί υπάρχει πρόβλημα τη διερμηνία. Μη με llega el español perfectamente, ε, δυστυχώς υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τους ε, διερμηνείς. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπάρχει ε, διερμηνία είναι δύσκολο να γίνει μία ακρόαση γιατί κατανοούμε μόνο οι ισπανόφωνοι. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε με την τελευταία σύνδεση για να δούμε εάν είναι λίγο καλύτερη. Γιατί διαφορετικά δεν θα γίνει άλλη σύνδεση. Ο κύριος ε, Ρομέρο έχει το λόγο. No, si no consigo la interpretación voy αν δεν τα καταφέρουμε με τη διερμηνία δεν, δεν θα μπορέσουμε, δεν θα το επιτρέψω δηλαδή, διότι αλλιώς παρακολουθούν μόνο οι Ισπανόφωνοι. Καλό σας απόγευμα, λέει η Πρόεδρος, δεν ξέρω αν με ακούτε καλά. Μάλιστα λέει ο Όποτε θέλετε να δούμε αν καταφέρομαι η δική σας σύνδεση να φτάσει θα το κάνω στα αγγλικά λέει ο μιλητής για να σας διευκολύνω για να δούμε διότι ήταν, προηγουμένως ήταν το πρόβλημα σύνδεσης ήχου λοιπόν πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποδεχθήκατε και όλους τους ε, πολίτες της Βενεζουέλας και τα μέλη της αποστολής Μου είναι αδύνατον, λέει ο μιλτής, να μιλήσω με τα ακουστικά διότι ακούω την επιστροφή. Μπορείτε να βγάλετε τα ακουστικά, λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζει ο προσκεκλημένος στα αγγλικά. Είμαι διευθυντής ε, ταμείου στην Βενεζουέλα, οργάνωσης που εκπροσωπεί θύματα αυθαίρετων ε, συλλήψεων στην Βενεζουέλα. Έχουμε πάνω από 200 δικηγόρους σε όλη την χώρα και πάνω από 1.500 ε, που, ακτιβιστές που συνεργάζονται μαζί μας. Θα ήθελα να αρχίσω με ένα παράδειγμα για να σας εξηγήσω πού βρίσκεται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Βενεζουέλα του Χεράρδο Καρέρο, ο οποίος κρατήθηκε στις 8 Μαΐου 2014 με άλλους 230 νέους. Οι άνθρωποι αυτοί ζητούσαν την απόλυση φοιτητών που κρατούνταν λόγω του ότι είχαν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις. Είχαν στήσει σκηνές μπροστά από τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στο Καράκας. Τους έβαλαν λοιπόν στη φυλακή και τους ανέκριναν και ο Θεράρδο κατήγγειλε ότι βασανίστηκε μαζί με άλλους. Τον Αύγουστο 2014 είπε ότι έδεσαν τα χέρια του αφού τα τύλιξαν πρώτα σε εφημερίδες για να μην κάνουν ουλές και τον κρέμασαν από έναν σωλήνα που πέναγε από το ταβάνι και έμεινε κρεμασμένος επί δύο ώρες. Τον χτύπησαν με ραβδιά πίσω από τα γόνατά του μέχρι που έσπασαν τα ραβδιά αυτά. Άφησαν δε μόλοπες στα πόδια του και στις κνήμες του και είχε και τους πόνες στην κοιλιά. Πόνες στην κοιλιά. Εμείς ως δικηγόροι Πήγαμε στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελία, για να καταγγείλουμε την κατάσταση αυτή και παρουσιαστήκαμε και στα δημόσια, στα ε, διεθνή μέσα επικοινωνίας και αναμέναμε ο Καρέρο ε, να φύγει από την φυλακή όπου βρισκόταν. Αντιθέτως όμως μεταφέρθηκε για έξι μήνες σε ένα κρύο απομονωμένο κελί χωρίς παράθυρα στο αρχηγείο της ε, αστυνομίας στο Καράκας χωρίς επισκέψεις, χωρίς επαφή με δικηγόρους, μέσα στο κελί του 24 χώρες, χωρίς φως. Η δε φυλακή του αποκαλείται τάφος και είναι και υπόγεια. Ακόμα υπάρχουν, κρατούνται άνθρωποι εκεί δεν έχουν καμία αίσθηση του χρόνου γιατί δεν φορούν και ρολόγια. Αυτή είναι η ιστορία του Χεράρδο Καρέρα, Καρέρο που έχει ανάγκη από ιατρική φροντίδα. Έξι μήνες μετά, όπως είπα, ο Χεράρδο μεταφέρθηκε πίσω στο μέρος όπου κατήγγειλε ότι είχε βασανιστεί. ακόμα δεν έχει λάβει την αναγκαία ιατρική φροντίδα και εξακολουθεί να υποφέρει από σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχει εκδορές στο δέρμα του και αποστήματα. Τα δόντια του έχουν πέσει και αναγκάστηκε να τα ξανακολλήσει με ε, κόλλα ο ίδιος μόνος του γιατί δεν ε, ε, λαμβάνει καμιά ιατρική φροντίδα. Υπάρχουν διακοπές στην σύνδεση που είναι υπερατλαντική, δυστυχώς με δορυφόρο και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, θα πολύ, είμαστε αναγκασμένοι να διακόψουμε. Ε, detainees, just as a result of demonstrations. We have registered 3,000 3,758 detentions. Sorry. Perdone, hay, ahora hay un problema de nuevo. Υπάρχει πάλι ένα πρόβλημα διότι δεν έχουν καλό ήχο οι διερμηνείς. Ε, άρα μπορείτε να φτάσετε στα συμπεράσματά σας είτε στα αγγλικά είτε στα ισπανικά διότι οι διερμηνείς δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν. We have registered 3,758 detentions from 2014. in total, 296 people uh, has been taken to jail by judicial orders. in it means between 40 days to one year. At this moment, there are 31 people in jail because... Επαναλαμβάνουμε. 77 άνθρωποι πολιτικοί κρατούμενοι το έπραξαν αυτό μεταξύ αυτών εμβληματικές φυσιογνωμίες όπως Λόπες και άλλοι αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι στις φυλακές υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έχουν σχέση με διαδηλώσεις όπως ο Γκονζάλες που έχουν, λέει, δημοσιεύσει επιθετικά μηνύματα Twitter ή προσβλητικά μηνύματα Twitter. Ας προσπαθήσω να ολοκληρώσω τώρα ε, λόγω χρόνου. Υπάρχουν περιπτώσεις φυλάκισης που είναι και ισοδύναμα με πολιτική κράτηση όπως απομόνωση με το, του, του Καρέρο που ανέφερα πριν περιορισμός ε, στις επαφές τους στην άμεση οικογένεια και στους δικηγόρους καθυστέρηση των δικαστικών διαδικασιών περίπτωση ενός δικηγόρου συνηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μαρσέλο Κροάτο δέκα χρόνια ε, όχι δέκα μήνες διορθώνει ο μιλητής πίσω από τα κάγκελα της φυλακής πάνω από ένα χρόνο τώρα κρατείται και κατοίκων και δεν έχει γίνει ούτε μία προκαταρκτική, προδικαστική μάλλον έρευνα σε βάρος του μέχρι τώρα. Χρησιμοποιούν τα, τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για να απαξιώσουν τους πολιτικούς αυτούς κρατουμένους παρακολουθούν με κοριούς και μικρόφωνα και δείχνουν τους ανθρώπους αυτούς και στα μέσα, κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μην σημαίνει τίποτα. Πάλι έχουμε προβλήματα διασύνδεσης με τη δορυφορική επικοινωνία.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 Σας ευχαριστώ κύριε Ρομέρο. Λυπάμαι γιατί υπήρχαν ε, τεχνικά προβλήματα, αλλά το μήνυμά σας πέρασε. Θα δώσω το λόγο στον τελευταίο προσκαλεσμένος μας, ε, προσκαλεσμένο μας ε, μέσω βίντεο link που δεν έχει και μεγάλη επιτυχία είναι ο κύριος Μαρίνο Αλβαράδο που είναι δικηγόρος της Προβέα του προγράμματος της Βενεζουέλας για την εκπαίδευση και τη δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να δούμε αν μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε. Hola. Hola. Hola. Με me, me ακούτε? Ναι. Θα πρέπει να μιλάτε πιο δυνατά για να μπορέσουμε να έχουμε διερμηνία στις διάφορες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να αρχίσετε, μιλώντας πιο δυνατά, δυνατά και αργά. Ο Είμαι ο Μαρίνο Αλβαράδο, εκπροσωπώ την Προβέα. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Ο κύριος Καμπρέρα σας μίλησε για τα θύματα που υπάρχουν στη Βενεζουέλα. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν, δεν είναι όλα αρνητικά ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα. Υπάρχουν και θετικά στον ε, τομέα, για παράδειγμα, της εκπαίδευσης. Επίσης έχουν ε, αυξηθεί οι εγγραφές στο Πανεπιστήμιο τα τελευταία έξι χρόνια. Επίσης, ε, οι αγροτικές οικογένειες έχουν περισσότερα αγροτεμάχια. Έχει γίνει καλύτερη διανομή. Υπάρχουν λοιπόν και κοινωνικές ε, αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Ως προς την ε, φτώχεια, Μέχρι το 2012 είχαμε μείωση του δίκτυ φτώχειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως μας απασχολεί το γεγονός ότι κατά το πρώτο έτος διακυβέρνησης του Νικολάς Μαντούρο η φτώχεια αυξήθηκε κατά 6% και όλοι οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι η φτώχεια αυξήθηκε από το 2014 και μετά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η διεθνής κοινότητα που ενδιαφέρεται για τη Βενεζουέλα στάθηκε σε αυτό το ζήτημα πρόσφατα. Τα θέματα κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα που ζήσαμε στη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια οδήγησαν σε πολλές κοινωνικές αναταραχές, ιδιαίτερα στους, πιο, στους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη ε, φτώχεια. Και βεβαίως είχαμε απεργίες κινητοποίησης, κλείσιμο ε, δρόμων μεταξύ των διαφόρων μορφών ε, διαδήλωσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι εργαζόμενοι της Βενεζουέλας έχουν αναλάβει τις διαδηλώσεις αυτές, τις δημόσιες αυτές ε, ε, διαμαρτυρίες. Η κυβερνητική απάντηση σε αυτούς τους κοινωνικούς κλειδονισμούς δεν ήταν δημοκρατικής υφής. Ε, κρίνονται ανατρεπτικές αυτές οι διαδηλώσεις και διώκονται οι διαδηλωτές. Ήδη πριν από τις ε, διαδηλώσεις του 2014 είχαμε περίπου 3.000 κρατούμενους, εκ των οποίων 150 ήταν συνδικαλιστές. Σήμερα 5.000 άνθρωποι στην ουσία διώκονται ποινικά. Πέρα λοιπόν από την ποινικοποίηση, στην ουσία καταστέλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με στόχο εκφοβισμού των ακτιβιστών. Δεν το επέτυχαν αυτό. Τίθεται ένα αμφιβόλο η νόμιμη διεθνής συνεργασία. Είχαμε μεγάλη βοήθεια και συνεργασία από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να βοηθήσουμε στην ενίσχυση της ε, δημοκρατίας. στην ουσία γίνονται απειλές, μάλλον οι εκπρόσωποι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δέχονται απειλές και θεωρούνται προδότες της πατρίδας. Στην ουσία χρησιμοποιούνται καθαρά κρατικά μέσα για να οδηγηθούν, για να διωχθούν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν είμαστε αντίθετοι στην κριτική. Θεωρούμε όμως ότι μπορεί κανείς να είναι υπέρ ή κατά της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά δεν μπορούν να διώκονται οι άνθρωποι αυτοί. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι για την δίωξη πολιτών. και για να αποδομηθεί η εργασία των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τα πιο φτωχά στρώματα της χώρας. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας στην ουσία έχει υποβαθμίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην ε, Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν γίνει καταγγελίες καθώς και στα διάφορα ε, θεσμικά όργανα όπως ε, τα Ηνωμένα Έθνη. Όμως δεν δέχονται τις επικρίσεις οι κυβερνητικοί και ούτε και τις συστάσεις και ε, δεν τηρούν τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, θεωρεί η κυβέρνηση ότι στην ουσία διώκεται η ίδια. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, όλες, ε, όλα τα φόρα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προβάλλουν ε, ένα ψευδές πλαίσιο αντίδρασης κατά της ε, Βενεζουέλας χωρίς να λάβουν υπόψη ότι δεν υπάρχει ε, δημοκρατία. Πρόκειται για ένα γεγονός που διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ανεπαρκής ε, αντιμετώπιση του ζητήματος. Και το δικαιοδοτικό ε, σκέλος δεν τηρεί τις αποφάσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υποβαθμίζεται η εργασία των ΜΚΟ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε να κάνουμε με ε, μια δημόσια εισαγγελία η οποία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα και γι' αυτό ακριβώς έχουμε ένα δίκτυο ατιμορρησίας στη χώρα της τάξης του 98%. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη δικαιοσύνης. Έχουμε να κάνουμε με μία δικαιοσύνη η οποία δεν μπορεί να εγγυηθεί μία δίκαια δίκη για όλους. Και στην ουσία το κράτος δεν κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει να ε, συνοψίσετε σας παρακαλώ. Θα ήθελα να αναφερθώ και στο σοφρονιστικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο προκαλεί τον θάνατο. Οι φυλακές της Βενεζουέλας είναι οι πλέον βίες στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν καταβληθεί προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις φυλακές, όμως το 2014, κύριοι βουλευτές, στις φυλακές είχαμε ανθρωποκτονίες και μεταξύ του 1999 και του 2014 είχαμε 6.472 ανθρωποκτονίες μέσα στις φυλακές. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί με ακούσατε. Εξ ονόματος των θυμάτων της ε, Γκουαρίμπα σας λέω ότι ευχαριστούμε γιατί μας εκπροσωπείτε για να καταπολεμήσουμε τις αδικίες και να υπάρχουν πραγματικές κυρώσεις κατά των υπευθύνων, όχι μόνο για τους θανάτους, αλλά και για τις ε, βίες διαδηλώσεις και τα βασανιστήρια που ζούμε συνεχώς. Σας ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος για τη συνεισφορά σας και για το συνεχιζόμενο αγώνα. Θα πάμε στις ε, ερωτήσεις των ε, μελών. Εγώ θα διατηρήσω εδώ στην έδρα, στο πάνελ, τα πρόσωπα που ήδη παρίστανται. Δεν θα μπορέσουμε όμως ε, για τεχνικούς λόγους να κάνουμε ερωτήσεις προς τους συνδεδεμένους με βίντεο link δυστυχώς. Έχουμε εδώ εκπροσώπους από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Έχουμε τα μέλη που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους ε, που έχουν άμεσο ενδιαφέρον στο θέμα. Ο κύριος ε, Ασής ε, που είναι πρόεδρος της Μερκοσούρ, ο κύριος Χαουρί, Ευρελάτ και ο Λουίς Ερνάντες ε, τις ε, κοινότητας των Άνδεων. Ο κύριος ε, Ασής. Θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι στόχος μας είναι να εποπτεύσουμε την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα σημεία της γης και υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Λατινικής Αμερικής. Έχουμε να κάνουμε βεβαίως με ένα κυρίαρχο κράτος, όταν μιλάμε για τη Βενεζουέλα, όμως επειδή ε, σεβόμαστε αυτή τη χώρα, γνωρίζουμε ότι η χώρα αυτή δεν έζησε υπό ένα δημοκρατικό καθεστώς πάντα. Θα πρέπει να δούμε θέματα τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στη Βενεζουέλα και δεν θέλουμε βεβαίως να υπάρχει παρεμβατισμός στα εσωτερικά της χώρας, στο εσωτερικό της χώρας. Και δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό που μας απασχολεί είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο κράτος αυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία χωρίς κράτος δικαίου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία χωρίς βασικές ελευθερίες από πολιτικής και πολιτιστικής πλευράς. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς όλα τα θύματα βίας, διότι εδώ δεν κάνουμε καμία διάκριση μεταξύ των θυμάτων, από όπου και αν προέρχονται. Πρόκειται για θύματα βίας και το σεβόμαστε αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κράτος δικαίου στη Βενεζουέλα και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μία διερεύνηση της όλης κατάστασης. Σήμερα έχουμε πολλές αμφιβολίες. Γιατί έχουμε να κάνουμε με πληθώρα περιπτώσεων όπου δεν τηρούνται τα δικαιώματα. Δυστυχώς το δικαιοδοτικό σύστημα δεν είναι ανεξάρτητο. Δεν υπάρχει ανεξαρτησία που θα πρέπει να χαρακτηρίζει ένα πραγματικό κράτος δικαίου. Έχουμε να κάνουμε με το δικαίωμα του συνέχεστε, της πληροφορίας, του εκφράζεστε. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με πληθώρα παραβιάσεων που μας αφηγήθηκαν ε, πολίτες που προέρχονται από όλο το φάσμα. Μιλάμε για το δικαίωμα του συνέχιστε, του εκφράζεστε και της ελευθερίας λόγου. Δυστυχώς σήμερα στη Βενεζουέλα υπάρχει μια τάση ποινικοποίηση της ελευθερίας του λόγου. Ε, υπάρχουν υπάρχει ε, πολιτική συνείδηση, αλλά η πολιτική συνείδηση και οι αντιρρησίες διώκονται. Δεν δικαιολογείται μια τέτοια κατάσταση. Δημοκρατία δεν σημαίνει καταπίεση της, ε, των μειονοτήτων. Δεν θα ήθελα να πω πολλά ακόμα, θα ήθελα να πω ότι ως επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας είχα έρθει σε επαφή με εκπροσώπους των αρχών της Βενεζουέλας. Εδώ και ένα μήνα ήταν αδύνατο να έρθω σε επαφή με τις διπλωματικές αρχές της Βενεζουέλας. Δεν ήθελα να έχουν καμία επαφή μαζί μας και δεν μπορώ να αποφανθώ γιατί συμβαίνει αυτό. Εμείς έχουμε μεγάλο σεβασμό για τη Βενεζουέλα, την ιστορία της, το λαό της και δεν θέλουμε να προβάλλουμε καμία παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εμείς μιλάμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα την οποία τιμάμε και αγαπάμε. Γιατί ξέρετε ότι είμαι Πορτογάλος και υπάρχει μια πολύ μεγάλη πορτογαλική κοινότητα στη Βενεζουέλα με την οποία έχουμε στενούς δεσμούς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Τεχάουρη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα συγχαρητήριά μου για την διοργάνωση αυτή και να προσθέσω και εγώ τη συμπάθειά μου, να εκφράσω τη συμπάθειά μου προς τα θύματα αυτής της ε, πολιτική στη Βενιζουέλα. Στην ε, συνεδρία της Ευρωλάτα ε, τις προηγούμενες ημέρες, Πρόεδρε, το συζητήσαμε εκτενώς το θέμα. Προφανώς με τους συναδέλφους από την Νότια Αμερική και πρέπει να σας ομολογήσω ότι είχαμε απόψεις αρκετά αποκλίνουσες. Η πλειοψηφία των Νοτιοαμερικανών θεωρούν ότι τα όσα λέμε και κάνουμε εδώ είναι παρέμβαση στα ιστορικά θέματα της Βενεζουέλας και ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τοποθετούμε μέσα. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελών του Ερωκού Κοινοβουλίου επαναλάβαμε μία άποψη και μία αρχή ότι μιλούμε πολύ συχνά για πράγματα που λαμβάνουν χώρα εκτός των συνόρων μας. Ίσως θα έπρεπε να μιλούμε ακόμα περισσότερο για τα όσα συμβαίνουν εντός. Αλλά το κάνουμε συνεχώς και για τη Βενεζουέλα και για άλλες χώρες του κόσμου. Ε, μιλούμε και θα μιλούμε όταν θεωρούμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως δεν πρόκειται για εσωτερική παρέμβαση. Είναι μια έκφραση αλληλεγγύης απέναντι στους πολίτες της ε, Βενεζουέλας. Είναι το ίδιο όταν μιλούμε για τους μετανάστες που έρχονται από τη Λιβύη και ασκούμε αυτοκριτική στις χώρες μας και πρέπει και μπορούμε να τοποθετούμαστε για τα τεκτενόμενα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όταν θεωρούμε ότι πλήττεται αυτή η παγκόσμια αρχή, η βασική αρχή σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ προσεγγίζω την όλη συζήτηση με τεράστιο σεβασμό και συμπάθεια προς, τους, προς τα θύματα. Εγώ μάλιστα είμαι αριστερός, είμαι σοσιαλιστής και επομένως υπό την έννοια αυτή ε, δεν μπορώ να κατανοήσω πώς η Ευρωπαϊκή Αριστερά ε, ε, κλείνει τα μάτια και θάβει το κεφάλι της δυνάμου απέναντι σε παραβιάσεις μιας θεωρητικά αριστερής κυβέρνησης. Εγώ θεωρώ ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το λέω στους συναδέλφους ε, πράττουμε, προχωρούμε σε μια πρακτική πόλωσης απέναντι σε τέτοια θέματα και δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή όταν βλέπουμε συμπεριφορές ε, επίκρισης προς τις κυβερνήσεις της Κολομβίας και του Μεξικού και γίνονται αυτά, τα κάνουμε αυτά αλλά είμαστε ανίκανοι να επικρίνουμε αντίστοιχα αριστερέ κυβερνήσει όταν προχωρούν σε αντίστοιχε παραβιάσεις. Εγώ είμαι λοιπόν αριστερός, είμαι σοσιαλιστής και θέλω και επιθυμώ να επικρίνω και να, να σημειώνω αντίστοιχε παραβιάσεις από όπου και να γίνονται αυτές. Δεν θέλω να είμαστε μονομεροί στην επίκρισή μας μόνο προς δεξιές κυβερνήσεις. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την αίθουσα και σε αυτό το όργανο πρέπει και μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί για τις παραβιάσεις αυτές και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην παράδοση και την ιστορία του Σοσιαλιστικού Κόμματος ε, της Ισπανίας. Στη δεκαετία του 20 μετά την επανάσταση στη Ρωσία, ε, κάποιος εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος πήγε στη Ρωσία για να καταλάβει αν εκείνη η επανάσταση που είχε μόλις ξεκινήσει ήταν μια επανάσταση που θα μπορούσε στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει η Ισπανική, το Ισπανικό ρεύμα. Ε, λεγόταν Φερνάντο Δελο Ρίος και ρώτησε τον Λένιν, ο Ρίος, εάν αυτό το κομμανιστικό κόμμα ήταν υπέρ της ελευθερίας. Και ο Λένιν του απήντησε σύμφωνα με την παράδοση ελευθερία για ποιο πράγμα. Και του είπε ο Ρίος ελευθερία για να είμαστε ελεύθεροι. Εγώ λοιπόν δεν κατανοώ πώς μπορεί μια κυβέρνηση της αριστεράς και αν ο κύριος ε, Τσάβες ή σήμερα ο κύριος Μαδούρο είναι αριστεροί, προχωρούν σε περιορισμό της ελευθερίας. Και εδώ είναι το σημείο, του, το, το κεντροπαρικό σημείο της συζήτησής μας. Είναι ο περιορισμός της ελευθερίας. Επομένως, ε, κυρίες και κύριοι, το συμπέρασμα μου είναι ότι τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο καιρό στη Βενεζουέλα είναι κινδυνεύουν σοβαρά να πλήξουν τη δημοκρατία αυτή και εμείς πρέπει να το πούμε για να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή, για να βοηθήσουμε το λαό της Βενεζουέλας, για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό το κάνουμε από αριστερή πλευρά και το κάνουμε από πλευρά και με πρόθεση φιλική προς τη Βενεζουέλα. Εφόσον λοιπόν τα πράγματα κυλούν στη Βενεζουέλα χωρίς ε, πολιτικούς κρατουμένους, χωρίς βία και μπορεί να τοποθετείτε και να εκφράζεται ο λαός, τότε όλα είναι καλά. Εγώ αυτά θα ήθελα να συμβαίνουν στη Βενεζουέλα. Εγώ ως πρόεδρος Ευρωλάτ αυτό το μήνυμα θέλω να διαβιβάσω. Ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές αρχές της δημοκρατίας χωρίς καμία ιδεολογική απόχρωση πρέπει να υπηρεσιούν πάντα δεν μπορούμε ως αριστερά να πλήττουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί τότε δεν είμαστε αριστερά πλέον. Και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Αριστερά να κλείνει τα μάτια της απέναντι σε μια λανθασμένη απεικόνηση, εξιστόρηση των γεγονότων, γιατί δεν το πιστεύει κανείς αυτό που μας λένε εδώ, ότι πρόκειται για κουντετά, για πραξικοπήματα που γίνονται συνεχώ. Έχουμε δει και τι καταστάσει ε, στην Αϊτή. Αν ήταν το πραξικόπημα που ήθελαν να κάνουν ε, στη Βενεζουέλα, τότε γιατί συναντήθηκαν εχθέ. Φτάνει με τα παραμύθια αυτά. Εμείς πρέπει να υπερασπιζόμαστε την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά είναι αυτά που εγώ πρεσβεύω. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Πρόεδρο πρόεδρος Χάουρη υπάρχουν διάφοροι που σα ε, επικροτούν σιωπηρά. Ο κύριο Δεγκράντε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ούτε σιωπηρά ούτε ανοιχτά χειροκρότησα, αλλά θα πω δημόσια ότι ταυτίζεται η θέση μου με τον πρόεδρο Χάουρη. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος αριστεράς βεβαίως, σε καμία περίπτωση, αλλά συμφωνώ με, τα, με τις εισαγωγικές τοποθετήσεις που ακούσαμε σήμερα εδώ. Η Επιτροπή του Κοινοβουλίου δεν επικρίνει ούτε την κυβέρνηση Μαδούρο, ούτε τη Βενεζουέλα, το κράτος της Βενεζουέλας, κάθε άλλο. Το κοινοβούλιο υπήρξε πάντοτε, προσέγγισε τα πράγματα με μεγάλο σεβασμό και μάλιστα με επιφύλαξη, αλλά επικρίνοντας κάποιες συμπεριφορές, συμπεριφορές που δεν ταυτίζονται δεν παραλληλίζονται με δημοκρατικά καθεστώτα, αλλά περισσότερο με απολυταρχικά καθεστώτα. Και αυτό το λέμε από διαφορετικές πολιτικές οπτικές γωνίες, προφανώς. Διότι είμαστε όλοι φίλοι της Βενεζουέλας και θα, και θα έλεγα έχουμε και συναισθήματα τουλάχιστον οι Ισπανόφωνοι εξημών προς τη χώρα αυτή. Γιατί όχι μόνο έχουμε επισκεφθεί τη χώρα αυτή, αλλά θέλουμε να ξαναπάμε. Και στην προσωπική μου διαδρομή, ε, εγώ μπορώ να σας πω ότι πολλές ιδέες έλαβα και input και βοήθεια από τη Βενεζουέλα, όταν στη δική μου χώρα δεν υπήρξαμε δημοκρατικοί και εκείνοι υπήρξαν. Τώρα, γιατί συνδέω την τοποθέτησή μου με τα λόγια του Πρόεδρου Χάουρη. Εγώ σε σχέση με τις ε, διάφορες ε, ανακοινώσεις της ελομελίας του Κοινοβουλίου που, έλεγε, που έλεγαν ότι το Κοινοβούλιο απέναντι σε αυτά τα γεγονότα όχι μόνο μπορεί αλλά πρέπει, πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Και θα έλεγα ότι έχουμε και απόλυτη νομική σαφήνεια, έχουμε το άρθρο 3 της συνθήκης της Ιδρυτικής που λέγει ότι σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές μας σχέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογραμμίζει τις βασικές αρχές και αξίες της και θα συνεισφέρει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτών με απόλυτο σεβασμό και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη χάρτα των ε, Ηνωμένων Αθνών. Ιδού λοιπόν και νομικά η νομιμοποίησή μας. Αλλά δεν είναι μόνο νομικό το θέμα. Έχουμε κάθε φυσικό δικαίωμα να το κάνουμε. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή το καθεστώς Μαδούρο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει στη φυλακή την αντιπολίτευσή του. Και ποιος μπορεί πλέον λογικά να αμφιβάλλει ότι χρησιμοποιεί δικαιολογίε για να μην επιτρέψει τη συμμετοχή στις εκλογές εκείνους που έχουν την επιθυμία και το δικαίωμα να εκπροσωπηθούν. Και, και εδώ μιλούμε για πολύ σημαντικό στοιχείο. Ε, φαίνεται ότι αναπτύσσεται πλέον ε, μία τάση από πλευράς του, λαού της Βενεζουέλας ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν τα πράγματα. Και δεν το λέει ο κύριος Ραμόν. Το λέμε εμείς, το λέμε οι φιλελεύθεροι, το λέει η κεντροαριστερά, η κεντροδεξιά, το λένε όλοι. Πρέπει να τοποθετούμαστε και να μιλούμε με καθαρή φωνή υπέρ των ιδεωδών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. πρέπει να πούμε στον κύριο Μαδούρο ότι δεν συμπεριφέρεται ως δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης, αλλά ως μονάρχης, ως εκπρόσωπος ενός απολυταρχικού καθεστώτος. Και ο λαός της Βενεζουέλας έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του με ελεύθερες, ελεύθερες και μη καθοδηγούμενες εκλογές. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε επίθετα και χαρακτηρισμούς, γιατί συμφωνούμε απολύτως, συμφωνούμε με το σεβασμό και τη φιλία που αισθανόμαστε προς τη χώρα αυτή, συμφωνούμε με τις αρχές που προκύπτουν και απορρέουν από την ιδρυτική μας συνθήκη και το κάνουμε από κάθε ιδεολογική τοποθέτηση. Όταν υπάρχει τέτοια ομοφωνία λοιπόν στο Κοινοβούλιο, κάποιο δίκαιο θα έχουν όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί. Ευχαριστούμε κύριε Δεγκράντες. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη εγώ πρόεδρε διότι δεν θέλω να επεκταθώ. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω και με τον κύριο Χάρου και τον κύριο Δεγκράντες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ομοφωνία και αυτή την κοινή εστίαση ιδιαίτερα επισημένοντας ότι εδώ δεν μιλούμε ούτε για αποκλήσεις ούτε για πολιτικές συνεννοήσεις. Στα ανθρώπινα δικαιώματα το ίδιο μας κάνει να γίνονται στο Μπουρούντι, στη Σαουδική Αραβία ή στη Βενεζουέλα αυτές οι παραβιάσεις. Επομένως, ορθώνουμε το ανάστημά μας για να υπερασπίσουμε τα, τα δικαιώματα των θυμάτων. Γιατί τα θύματα προέχουν. Είναι πιο σημαντικά από κάθε άλλο πράγμα και πολιτική προσέγγιση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συνεργάτες ε, και συνεισφέροντες ε, σε αυτήν τη συναδρίαση και για την καθημερινή τους προσπάθεια και δουλειά τους. Γιατί ήταν εκεί από πριν, συνεχίζουν να αγωνίζονται και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται. Και πρέπει να επιτηρούμε ότι όλα αυτά θα είναι αποτελεσματικά και θα οδηγήσουν σε δικαιώματα. Λοιπόν, έχω 4-5 ακόμα... 4-5 ε, μέλη που ζητάνε το λόγο και μετά θα ήθελα τα μέλη του πάνελ να απαντήσουν για να έχουμε λίγο ακόμα περιθωρία. Ο κύριος Χένκελ παρακαλώ. Δυστυχώς τα όσα συμβαίνουν τώρα να μιλήσω και αγγλικά θέλετε τα όσα συμβαίνουν συνεχίζω στα αγγλικά Δυστυχώ είναι χαρακτηριστικά και για ορισμένε άλλε χώρες της ε, Νότια Αμερικής. 50 και παραπάνω χρόνια καταπίεση στην Κούβα, για παράδειγμα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διεξαχθεί προεβδομάδων συζήτηση σχετικά με κάποιες πολύ δυσάρεστες τάσεις που σημειώνονται στην Ουγγαρία. Βρήκα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι άλλοι πρόεδροι κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων άρχισαν να γύρουν την φωνή τους για να εκφράσουν τις, τις ανησυχίες τους για το τι σημαίνει στην Ουγγαρία. Κάτι που μου λείπει ωστόσο για την Νότια Αμερική. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και απέναντι στις άλλες κυβερνήσεις. Αυτό που μου φαίνεται να λείπει για την Νότια Αμερική είναι οι κριτικές απέναντι για παράδειγμα στη κυβέρνηση χιλής της Βραζιλίας αυτές που γίνονται και απέναντι στη Βενεζουέλα. Αυτό για μένα είναι και εκπληκτικό αλλά και ε, αποθαρρυντικό. Θα πρέπει όταν συναντούμε πρόσωπα από άλλες δημοκρατικές κυβερνήσεις της Νότιας Αμερικής θα πρέπει να τις ενθαρρύνουμε να επικρίνουν οι ίδιες την Βενεζουέλα, την κυβέρνηση Βενεζουέλας, να μην περιμένουμε μόνο από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να καταδικάζουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα εκείνη. Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ, να σας συγχωρώ για την διοργάνωση αυτής της συνάντησης, γιατί έχει σημασία να δούμε τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα. Θα ήθελα να σας πω για το εξής. Πριν μπω στην πολιτική, ε, εδώ και 20 χρόνια ε, δούλευα σε ΜΚΟ, στη χώρα μου και αλλού. Και θα πρέπει να πω ότι όταν γίνεται λόγος για την Επιτροπή των Θυμάτων της Γουαρίμπα και του Γκόλπε Κοντινουάδο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πρόκειται για μία ΜΚΟ γιατί η πολιτική εμπεριέχεται ε, στην ονομασία της οργάνωσης. Ε, λυπούμε γιατί όταν υπάρχει βία υπάρχουν θύματα από όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα αθώα ε, ε θύματα, αλλά τα λόγια της, ε, του κυρίου Καμπρέρα δεν με έπεισαν γιατί φαίνεται ότι εργάζεται για για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, αλλά εγώ ποτέ δεν δούλεψα για την κυβέρνηση όταν ήμουν σε μία μήκη όπως η κυρία Καμπρέρα. Ε, έχω μία ερώτηση, γιατί λυπάμαι για το γεγονός ότι στη Eurolat δεν έχουμε κοινή δήλωση από τους πολιτικούς και αναρωτιέμαι πού έγκυται η αλληλεγγύη της κοινωνίας των πολιτών ως προς τη Λατινική Αμερική, που έγκυται η στήριξη δηλαδή στις οργανώσεις της Βενεζουέλας. Τι γίνεται με τους δημοσιογράφους, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σε διεθνές επίπεδο Υπάρχει ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται και σε επίπεδο Λατινικής Αμερικής. Ο κύριος Κόουσο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεγκράντες είπε είπε ακριβώς ε, για την πεμπτουσία της δημοκρατίας και συμφώνω μαζί του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι περίεργη η εκπροσώψη. Έχουμε μία μήκυο η οποία σχετίζεται με κόμματα της αντιπολίτευσης. Εδώ μία κυρία που ανήκει σε μία ε, ε, πολιτική οργάνωση της αντιπολίτευσης, αλλά έχουμε και να κάνουμε και με έναν πολιτικό, ο οποίος ήταν αναπόσπαστο ε, μέρος ε, της ε, κυβερνητικής πολιτικής. Νομίζω ότι θα, πρά... θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είχαμε μία εκπρόσωπο των θυμάτων. Έγινε λόγος για τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Περίεργο γιατί η Επιτροπή αυτή είχε στην ουσία συνεδριάσει και στην χιλή του Πινοτσέτ, υπό την αιγίδα μίας οργάνωσης του Πινοτσέτ. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε παρά το ότι πρόκειται για ε, υποχρεώσεις και δικαιώματα τα οποία σχετίζονται με Κυβερνητικέ και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κύριε Χάουιτ, δεν ε, σα τρέφω μεγάλο συμβασμό, αλλά δεν ε, συμφωνώ μαζί σα. Έχουμε 7 ψηφίσματα τα τελευταία χρόνια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση με άλλες χώρες. Μιλάμε για ελεύθερες ε, εκλογές. Και έχασε τις εκλογές. Ε, ο προκάτοχος κάτι το οποίο το δέχτηκε. Είναι πολύ ε, φυσικά αρνητικό το ότι ο προκάτοχος δεν δέχτηκε να γίνει λόγος για αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε ε, για βία θα πρέπει να λάβετε υπόψη την ε, χώρα της Ονδούρας. Δηλαδή στο Μεξικό έχουμε 86 δημοσιογράφους που ε, δολοφονήθηκαν και στη συνέχεια να δούμε την Κολομβία με 55%. Μιλάμε για, δημοσιογρα... για τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα. Γιατί να μην μιλάμε για το Σαλβαδόρ, την Κολομβία και τη σονδούρας και να μην ε, μιλάμε για να μην μιλάμε κατά αυτών των οργανώσεων. Τι περίεργο, όταν ε, η αριστερά κερδίζει τότε μιλάμε για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας λαστάσουμε στη Βενεζουέλα. Από το 1999 η φτώχεια από το 49% έφτασε στο 27%. Μιλάμε για την απόλυτη ένδυα. Και αυτό το δέχτηκε και η UNESCO και η ΦΑΟ. Μιλάμε για ένα 17% αρχικά και 7% στη συνέχεια. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και οι υπηρεσίες υγείας έχουν πολύ βελτιωθεί. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο κύριος Χάουρη μίλησε για ατιμορρησία. Μιλάμε για 40.000 αγνοούμενους στο Μεξικό. Τιμορρησία 100%. Και εδώ μιλάμε ε, για 43 φοιτητές που ε, βασανίστηκαν. Μιλάμε για καταστολή. Ας δούμε τι γίνεται με την ε, πολιτοφυλακή στις ΗΠΑ που πρόκειται για ε, ένα καθαρά στρατιωτικό ε, σχήμα. Δηλαδή, ό,τι ισχύει για τη ΣΥΠΑ δεν ισχύει στη Βενεζουέλα. Εδώ μιλάμε για ε, φοιτητές μέσα σε εισαγωγικά με όπλα και οβίδες. Στη χώρα μου όταν είχαμε οβίδες και όπλα δεν δεχόμασταν να πούμε ότι υπήρχαν, ε, υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση στην ε, χώρα μου. Δεν θα το δεχόμαστε αυτό ως προς τη δικαιοσύνη και με αυτό τελειώνω. Κρατούμενοι. Γιατί τα αστυνομικά στοιχεία μιλάνε από μόνο τους. Μιλάμε για 43 δολοφονίες από αστυνομικούς. Αυτό το λέει και η κυβέρνηση. Οι 35 από την αντιπολίτευση. Εννέα αστυνομικοί μεταξύ αυτών, αστυνομικοί που υπηρετούν τη χώρα. Ο δημόσιος κατήγορος μίλησε για 215 πράξεις και σε 13 περιπτώσεις έγινε δίωξη. Έχουμε ακόμα 21 περιπτώσεις που διερφωνούνται. Ε, δύο περιπτώσεις ανθρωποκτονίας, ε, τρεις ε, περιπτώσεις στη Μέριτα και μιλήσαμε και για επτά θανάτους, αλλά σε μία περίπτωση μιλάμε για ένα μικρό παιδί το οποίο σκοτώθηκε. Ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν για τιμωρησία γιατί διώχθηκαν οι υπεύθυνοι. Δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν μιλάμε για τιμωρησία. Ευχαριστούμε για τον κύριο Κόουσο. Τώρα, πέρα από τους ε, προσκεκλημένους, όλοι αξίζουν το σεβασμό μας εδώ. Όλοι και τα μέλη και οι προσκεκλημένοι μας και δεν χρειάζεται να κατηγορούμε κανέναν. Για την εκπροσώπηση θα απαντήσω μόνο για την υποχρέωσή μου. Είναι οι πολιτικέ ομάδε που πρότειναν του συμμετέχοντες. Η κυρία Σολορθάνο την πρότεινε η ομάδα σοσιαλιστών, η κυρία Καμπρέρα, η δική σας ομάδα, ο κύριος Ρομέρο από τους Φιλελεύθερου, ο κύριος Αβελέδο από το ΕΛΚ και ο κύριος Αλβαράδο με τον οποίο μιλήσαμε μέσω βιντεολίνκ των Πρασίνων. Δηλαδή, οι πολιτικέ ομάδες, σε πάση περιπτώσει, υπέβαλαν τις προτάσεις τους. Εμείς απλώς επιβεβαιώσαμε ότι πρόκειται για φορείς και οργανώσει που όντως δραστηριοποιούνται και σε ό,τι με αφορά προσωπικά, εγώ ασχολήθηκα η πρεσβεία να ενημερωθεί εγκαίρω και να έχει προσκληθεί επίσης εγκαίρω. Και μάλιστα επέμεινα στι τελευταίε μέρε να στείλει εκπρόσωπο προσπάθησα να έρθω σε επαφή με τον πρέσβη χωρίς επιτυχία. Είναι ο, πρός, ο πρώτος πρέσβης τον οποίο δεν καταφέρω να μιλήσω να σας πω. Εν πάση τόσο τους προσκαλέσαμε και εκείνοι έκριναν ότι δεν έπρεπε να έρθουν, ότι δεν άξιζε. Τώρα, και εγώ ήθελα τα πράγματα να είναι πιο ισορρόπα, γι' αυτό προσεκάλεσα και την πρεσβεία. Και αυτό κάνουμε πάντοτε σε αντίστοιχες περιπτώσεις Προσπαθούμε δηλαδή η συζήτηση να είναι δημοκρατική, ανοιχτή και ισορροπημένη στο μέτρο του δυνατού. Η πρεσβεία όμως ε, δεν είναι θέληση, το οποίο ήταν έκπληξη για τα μέλη της Επιτροπής μας, γιατί συνήθως οι διπλωματές συμμετέχουν. Και βεβαίως το ίδιο κάναμε και για το Μαξικό και σήμερα και αύριο θα, το, θα κάνουμε το ίδιο για την ε, ε Λωρίδα της Γάζας, για την Ουκρανία η λειτουργία της Επιτροπής είναι να επιτηρεί και να υπερασπίζεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η λειτουργία και εγώ ως πρόεδρος αυτό θα κάνω. Μόνο, μόνο το εξής, να σας ευχαριστήσω για την εξήγηση. Εγώ δεν ήθελα καθόλου να κατηγορήσω κανέναν, απλώς ήθελα να επισημάνω ε, ένα γεγονός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω πού είδατε αυτά τα νέα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, έχετε την κασέτα που ακούμε και από την πρώην Σοβιετική Ένωση και τη βάζετε συνέχεια. Νομίζω ότι δεν, ε, δεν με τιμάτε και στην ουσία είναι δηλητηριώδη τα βέλη σας, χωρίς λόγο. Βλέπω ότι, ε, ότι, ότι ότι ακούτε την ίδια, βάζετε την ίδια κασέτα μπροστά και μου θυμίζει σαν να πρόκειτο ε, εσείς, εσείς δεν τιμάτε τη διοργάνωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Ραμόν Αβελέδο, τον κύριο Τέρο που είναι εδώ, ε, τον κύριο Μπετενκούρ, όλους τους ε, Ισπανόφωνους και θα ήθελα να πω στο φίλο μου Ραμόν ευτυχώς που είμαι ε, φιλελεύθερος. Διαφορετικά ποιος ξέρει τι δηλητηριώδη βέλη θα έριχνα και εγώ, όπως ο προλαλή σας. Ξέρουμε ότι ο λαός της ε, Βενεζουέλας ε, πλήττεται, έχει θυματοποιηθεί και δεν μπορούμε να πούμε ότι τίποτα δεν του συμβαίνει. Είναι ένας θαραλέος λαός και θα πρέπει να τον ε, τιμάμε. Δεν ξέρω αν θα είχα το θάρρος να βρίσκομαι εδώ υπό αυτή την ιδιότητα. Δεν θα ήθελα να κάνω δηλώσεις καλών προθέσεων. Νομίζω ότι η συζήτηση έχει πολιτικοποιηθεί ιδιαίτερα. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά υπάρχουν, ε, υπάρχει ατιμορρησία, υπάρχουν αυθαίρετες αποφάσεις, υπάρχει ε, μία, ένας παρεμβατισμός της εκτελεστικής εξουσίας τη δικαιοδοτική και ούτω καθεξής. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, δεν υπάρχει ελευθερία του εκφράζεστε, αλλά μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των πολιτών πρωτίστως. Και επειδή είμαι Πορτογάλος, όπως και ο συνάδελφος ε, δίπλα μου, έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινότητα Πορτογάλων στη Βενεζουέλα. Είναι και αυτοί οι θύμα της κατάστασης, ζουν αυτή την κατάσταση. Όταν εγκαταστάθηκαν εκεί προσπάθησαν να βρουν την τύχη τους σε μια άλλη χώρα όπου να μπορέσουν να ευημερούν, να δημιουργήσουν, να συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας χώρας ε, ευημερίας. Αλλά δυστυχώς ζουν τις ε, δολοφονίες, την ε, δίωξη των ε, θυμάτων και μας τα αναφέρουν όλα αυτά. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και θα πρέπει να επιβάλλουμε στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εδώ έχουμε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και θα ήθελα να πω τι μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση. Είναι ενωμένη. Γιατί στις προσεχείς εκλογές θέλουμε να υπάρχει μία εναλλακτική για την ανάληψη της εξουσίας. Είναι πραγματικά ενωμένη η αντιπολίτευση. Γιατί θα πρέπει να τύχετε ευρύτερη υποστήριξη ή δυνατόν. Όπως είπε και ο Ραμόν, πώς εμείς οι Ευρωπαίοι μπορούμε να σας βοηθήσουμε τη στιγμή που είναι διχασμένη η Λατινική Αμερική και δεν ε, σας υποστηρίζει. Μιλήσαμε για τις διασκέψεις της Eurolat και η Ελάκ προσπάθησε να συνεισφέρει, αλλά δεν μας το επέτρεψε η Λατινική Αμερική γιατί θεώρησε ότι υπάρχει παρέμβαση, παρεμβατισμός στα εσωτερικά των χωρών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Θούβερ. Θα μιλήσω και εγώ πορτογαλικά, λέει η κυρία Ζούμπερ. Νομίζω ότι γίνεται μία μεγάλη σύγχυση μεταξύ του νομίμου δικαιώματος να ε, αναρωτιόμαστε για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ε, ιδεολογημάτων του καθενός. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τους προσκαλεσμένους που αντικατοπτρίζει φυσικά και την πλειοψηφία της τάσης του Κοινοβουλίου έναντι της Βενεζουέλας. Πρόκειται για μια ισορροπία που αντικατοπτρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν με σοκάρει δηλαδή το γεγονός καθε αυτό. Αλλά η πρώτη παρεμβαίνουσα μίλησε για ορισμένα γεγονότα και οι άλλοι παρεμβαίνοντες ε, πέρα από γεγονότα άρχισαν να γνωμοδοτούν για τη διακυβέρνηση, για την οικονομία, για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, για τη φτώχεια, για τη λιμοκτονία και για όλα τα συναφή. Αυτά δεν είχαν σχέση με το θέμα υποσυζήτηση. Γιατί όλοι έχουμε γνώμη αλλά δεν θα κρίνουμε εμείς ποια είναι η πολιτική πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει η Βενεζουέλα. Το αποφάσισε ο λαός της Βενεζουέλας αυτό και δεν μας πέφτει λόγος. Εκλογές που διενεργήθηκαν ε, με την παρουσία διεθνών παρατηρητών. Υπόθηκε ότι θα πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη. Εμείς, η ομάδα μας, αντιτάχθηκε σε αυτές τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτον, γιατί υπάρχει πολιτική χειραγώγηση και αυτό συμβαίνει πάντα προεκλογικά. Αυτό αποτελεί παράδοση. Λέμε ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Για να είναι ανεξάρτητη και αποτελεσματική, δεν θα πρέπει να δέχεται αυτές τις πιέσεις και τις παρεμβάσεις ως προς το διαχωρισμό των εξουσιών. Θεωρούμε ότι οι περιφερειακοί οργανισμοί της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής εποπτεύουν την κατάσταση. Στην ε, τελευταία συνεδρίαση της ε, Eurolat προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε μια συνένεση αλλά εκπροσωπούνται, εκπροσωπείται όλο το πολιτικό φάσμα, γιατί μιλάμε για, συνιστόσα, για τη συνιστόσα της Λατινικής Αμερικής, η οποία απαρτίζεται από πολλές πολιτικές τάσεις. Επίσης έγινε λόγος για την ε, παρέμβαση της ε, Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδώ Μιλάμε για δεδομένα τα οποία ε, δεν δέχονται πολλές χώρες, όχι μόνο η Βενεζουέλα. Εμείς απορρίπτουμε απόλυτα αυτή τη χειραγώγηση της ακρόασης με άλλους στόχους, γιατί υπάρχει σκοπιμότητα και δεν είναι τυχαίο ότι δεν γίνεται λόγο για το πραξικόπημα του 2002 στη Βενεζουέλα. Θα πρέπει να φτάσετε στα συμπεράσματά σας χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. που νομιμοποίησε μια κυβέρνηση που ε, αναγνώρισαν οι ΙΠΑ και η Ισπανία, αλλά το BBC και το Άρτε μίλησαν για αυτό το πραξικόπημα του 2002 και είδαμε ότι αλλιώς είχαν τα πράγματα στη Βενεζουέλα. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους. Ε, πρώτα στην κυρία Καβρέρα για κάποια συμπεράσματα και απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου έγιναν. Για τον κύριο Ασής που μας ρώτησε για τη δικαιοσύνη. Εμείς συναντηθήκαμε με το Υπουργείο, με τους υπευθύνου και παρακολουθήσαμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Υποβάλαμε ερωτήσεις, είχαμε και καταδικαστικές αποφάσεις συγκεκριμένες από τα δικαστήρια. Και ναι, εγώ ε, είμαι εκπρόσωπος του Υπουργείου ε, που είναι υπεύθυνο για θέματα κατοικίας και ως εκπρόσωπος του Δημοσίου ε, αυτό δεν μου αφαιρεί το δικαίωμα να απαιτώ την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα αυτά. Μπορώ λοιπόν να συνεχίσω να αγωνίζομαι ακόμα και εκπροσωπώντας το δημόσιο. Τώρα αναφερθήκατε στους ε, σπουδαστές, στους φοιτητές που κρατούνται ότι υπέστησαν ε, βασανιστήρια κτλ. Ο κυρίος Όσκα έχασε το χέρι του επειδή του πέταξαν υποτίθεται κάποιοι ειρηνικά διαμαρτυρόμενοι φοιτητέ ε, εκρηκτικά. Υπήρξαν θύματα, νεκροί. Έχουμε δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν σφαίρες της μοντελικής στήλη και έχουν μείνει παράλληλοι για πάντα. Έχουμε συναδέλφους που χτυπήθηκαν και έπαθαν σοβαρές σωματικέ βλάβες από αυτές τις ε, οργανώσεις των ειρηνικών διαδηλωτών. Δείτε τις περιπτώσεις, δείτε τι έχουν πάθει. Όταν μας λέτε ότι έχουμε φοιτητές, ειρηνικούς φοιτητές που διαδήλωναν και τους κρατούμε στις φυλακίες. Πρέπει να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη στη χώρα και ποια είναι τα θύματα. Και να σας θυμίσω ή να σας πληροφορήσω ότι το 2013 η Επιτροπή μας συνένωσε και τις οικογένειες των θυμάτων του 2013 του πραξικοπήματος εκείνου όπου είχαμε υποψήφιο ο οποίος όταν είδε ότι τα αποτελέσματα ήταν δεν ήταν καλά για τον ίδιο, κάλεσε όλους τους οπαδούς του σε βίαιες διαδηλώσεις. Αυτό συνέβη. Και οι ομάδες αυτές επετέθησαν σε κέντρα υγείας, σε εκλογικά κέντρα. Δεν τους ενδιέφερε ότι μέσα υπήρχαν άνθρωποι και είχαμε θύματα. Είχαμε τρία μικρά παιδιά που πέθαναν, έχασαν τη ζωή τους στα επεισόδια εκείνα. Ένας πολιτικός λοιπόν ηγέτης κάλεσε σε βίαιο ξεσηκωμό τους οπαδούς του. Αυτό συνέβη. Σας ευχαριστούμε κυρία Καβερέρα. Ο κύριος Αβελίδο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη για τη συνεισφορά τους. Ο καθένας έχει δικαίωμα και είναι τιμή του να εκφράζει την απόψή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και στα Εθνικά βεβαίως Κοινοβούλια. Αλλά στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας δεν είναι έτσι. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου εκεί θεωρεί ότι είναι η ιδιοκτησία του η αίθουσα. Και δίνει το λόγο ή δεν το δίνει όπως νομίζει. Και έχουμε μέλη του Κοινοβουλίου που έχουν απομακρυνθεί επειδή εξέφρασαν την πολιτική τους άποψη χωρίς άλλη διαδικασία, χωρίς συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Χωρίς τίποτα από αυτά. Και με κάθε σεβασμό λέω ότι υπάρχουν κάποιες ιδεολογικές τάσεις. Υπάρχει μια ταυτοποίηση με ορισμένες θέσεις και θεωρούν ότι όλα αυτά που λένε και κάνουν είναι ιερά και όλα τα υπόλοιπα είναι απλά απόψεις. Και έτσι η εξήγησή τους είναι κάπως ε, ταυτόσιμη λέγοντας ότι είναι έτσι επειδή εγώ έτσι το λέω. Αλλά δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Δεν εξηγούνται έτσι τα πράγματα. Τώρα θα προσπαθήσω να μείνω στον χρόνο μου δίνεται σεβόμενος όλους τους ομιλητές λέγοντας τα εξή. Καταρχά. εμείς είμαστε υπέρ μιας Βενεζουέλας όπου μπορούν να μπορούν να ειρηνικά να συνυπάρξουν όλοι οι πολίτες με όλες τις πολιτικές προτιμήσεις χωρίς διακρίσεις. Η βία που είχαμε τα τελευταία χρόνια που είναι καταδικαστή όποιος είναι να προκύπτει από το γεγονό ότι στη Βενεζουέλα οι θεσμοί, τα θεσμικά όργανα, τα υπουργεία, η δικαιοσύνη, όλα αυτά κυριαρχούνται από μια πολιτική προσέγγιση από την κυβέρνηση στην ουσία. Γιατί το Σύνταγμα λέγει ότι οι δικαστές θα πρέπει να ορίζονται βάσει διαγωνισμού. Αλλά δεν γίνεται έτσι στην πράξη ότι χρειαζόμαστε ειδική πλειοψηφία για να ορίζουμε τους ε, υψηλούς δικαστικούς λειτουργούς, τους εισαγγελείς κτλ. Αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική ενισχυμένη δηλαδή πλειοψηφία, αλλά απλή πλειοψηφία. Για να οριστούν απλά δημόσιοι υπάλληλοι φιλικά κείμενοι προς την κυβέρνηση, οι οποίοι δεν έχουν καμία άλλη κατάρτιση για τέτοιου είδους θόκους. και για την ε, συνάδελφο που μιλάει εξ ονόματος Επιτροπής των Θυμάτων και αυτή θα πρέπει να διοικείται από ένα αντικειμενικό πρόσωπο και όχι πρόσωπο που έχει ορίσει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, όπως συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Χρειαζόμαστε δικαιοσύνη για όλους λοιπόν, αληθινή δικαιοσύνη. Και το έλλειμμα της δικαιοσύνης που έχουμε στη Βενεζουέλα είναι ακριβώς αυτό. Έχουμε ένα θέμα αξιοπιστία των θεσμών. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και κάποια στιγμή βεβαίω θα αλλάξουν αυτά. Γιατί τι αρέσκεται η κυβέρνηση να λέγει ότι η χώρα άλλαξε για πάντα, ότι ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι όλες οι πλειοψηφίες, δεν είναι, καμία μάλλον πλειοψηφία δεν είναι αιώνια. Και τα πράγματα αλλάζουν μία μέρα κάποιο είναι πλειοψηφία, την άλλη είναι μειοψηφία. Κάποιο λέει κάτι εκτό μικροφώνου. Μάλιστα, βεβαίω έχετε δίκιο, λέει ο μιλητή. Η πρόεδρο λέει: Αν μπορείτε, αν θέλετε να μιλήσετε χωρί μικρόφωνο, αν θέλετε να πάρετε για λίγα δευτερόλεπτα. Ε, ζητώ συγγνώμη, πρόεδρε, αλλά πραγματικά. Ε, πραγματικά ε, ήθελα να αντιδράσω προς αυτά που ακούω γιατί μου φαίνονται επανέρχεται ο μιλητή και λέει εγώ συμφωνώ απολύτω μαζί σα. τα πράγματα πρέπει να γίνονται βάσει της ψήφου δημοκρατικά Δηλαδή αυτό που θα επιλέγει η πλειοψηφία. Αυτό είναι το ορθό, αυτό είναι το σωστό. Προχωρώ. Στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας μάλλον δεν αποδέχεται η κυβέρνηση ότι να τοποθετείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, το θεωρεί αυτό παρέμβαση στα εσωτερικά θέματα. Ενώ άλλα κοινοβουλία του κόσμου έχουν τοποθετηθεί. Προφανώ βέβαια το δέχονται όταν είναι ευνοϊκέ οι τοποθετήσει. Αλλά σιωπή σε σχέση με άλλε τοποθετήσει άλλων κοινοβουλίων. Η γερουσία τη Ουρουάη, προσέξτε, η, της Κολομβίας, το Κογκρέσο του Περού, η, η αίθουσα της Χιλής, η γερουσία της Βραζιλίας, της Κωνσταντίνα, όλες αυτές οι αίθουσες των κοινοβουλίων σημείωσαν τα ίδια συμπλήν λέει ο ομιλητής, αλλά σιωπά η κυβέρνηση Βενεζουέλα απέναντι σε όλα αυτά, γιατί θέλει όλα αυτά να τα παρουσιάζει ω απεικιοκρατική αντιμετώπιση των Ευρωπαίων. Όμω υπάρχουν αξίε Τη δημοκρατίας που είναι παγκόσμιες και συνολικές, καθολικέ με συγχωρείτε. Και δεν μπορεί κάποιο να μένει μονοπωλιακά στο ένα, σε μία ερμηνεία, τη δική του ερμηνεία των πραγμάτων. Αυτό δεν το καταλαβαίνει η κυβέρνηση Βενεζουέλας. Ο κύριο Κόουσο, για παράδειγμα, ξαφνιάζεται που ε, αναφέρομαι στην Επιτροπή των, ε, της, των Κοινοβουλίων της Νοτιού Αμερικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό προκύπτει από την ίδια συνθήκη όμως. Από την ίδια Διεθνή Συμφωνία. Τη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Νοτιού Αμερικής. Γιατί απεσύρθη η Ουρουγουάη, γιατί απεσύρθη η Χιλή, γιατί η Βραζιλία εφόσον είναι ένα ε, όργανο και μέσω των Ηνωμένων, των Πολιτείων όπως λέτε εσείς γιατί δεν απεχώρησαν. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για κυβερνήσει που είναι επικριτικέ της Αμερικανικής. Όπως και η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα ποτέ δεν υπήρξε, λέει ο μιλητής, ποτέ, ποτέ δεν υπήρξε υπηρέτη των Αμερικανικών συμφερόντων. Ε, υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις. Όπως στη σύνοδο της Πούντα Ελέστε, όταν, κατηγο... όταν ε, δώσαμε την... Ε, ε, ο, ο, ο πρόεδρος Τσάβες είπε για την εισβολή στη Δομινικανή Δημοκρατία, το είπε ο Ισπανός Βασιλιάς, γιατί δεν το βουλώνεις όπως θυμόμαστε όλοι. Εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Αλβαράδο όπως και οι υπόλοιποι εξέφρασαν την άποψή τους. Υπογραμμίζοντας πτυχές ενδεχομένως που εγώ δεν θα, δεν θα επέλεγα. Αλλά Είχαμε κυβερνήσει και πριν το 98 και μετά το 98. Ο καθένα έχει δικαίωμα στην απόψη του. Έχει μια ζυγαριά, μια δική του ερμηνεία των πραγμάτων. Θυμάμαι ένα φιλμ που είχε βγει πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν φοιτητή που λεγόταν. Il Vivant του Κώστα Γαβρά. Τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ισπανόφωνοι μπορούσαν να το δουν εκείνο, την εποχή εκείνη, διότι ε, το είχαν αποκλείσει βεβαίω. Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία του φίλου του. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε ε, πολιτικούς ε, πρόσφυγες και ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί σε άλλες χώρε λόγω των πολιτικών του πεπιθήσεων. Ο Φερνάντο Ρίος, για παράδειγμα, μεταξύ αυτών. Ο Αγούστο Πισουνιέρ. Είχαμε την ευκαιρία, την ευτυχία, να έχουμε την ε, στήριξη συγκεκριμένων ανθρώπων και φίλων. Άρα λοιπόν πιστεύουμε τα μεγέθη των Εθνών όταν μας δίνουν στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη των δικτών της στόχιας ή όχι. Ή του ΦΑΟ που προκύπτουν από τα Ηνωμένα Αθήνη. Έθνη. Πρέπει να επικαιροποιήσουμε τα μεγέθη. Και όσο επικαιροποιούνται τα μεγέθη προκύπτει ότι εάν υποχώρησαν κάποια μεγέθη λόγω της υπερβολικής αύξησης του πληθωρισμού προηγουμένω, τώρα γίνεται το αντίστροφο. Είμαστε πιο φτωχοί στη Βενεζουέλα τώρα παρά πριν από 15 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν όμως οι οργανισμοί των ΗΕ λένε πράγματα που μας πάνε καλά από πλευράς κυβέρνησης, οκ. Όταν αναφέρονται σε βασανιστήρια ή άλλες ε, παραβιάσεις τότε δεν θέλουμε να τα ακούμε αυτό. Και αυτό που ήθελα επίσης να τονίσω είναι το επιχείρημα σχετικά με την παρέμβαση στα ιστορικά πράγματα της Βενεζουέλας. Όταν από το εξωτερικό δηλαδή έχουμε επικρίσεις. Τότε λέει η κυβέρνηση αυτό είναι παρέμβαση. Και εμείς είμαστε ανεξάρτητοι και δεν δεχόμαστε παρεμβάσεις. Και θυμάμαι όταν συζητούσαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Χιλή και στην Κούβα, εκεί είχαμε να κάνουμε δικτατορίες και αυτή ήταν η μόνιμη απάντησή τους οι δημοκρατίες δέχονται τις επικρίσεις της διεθνούς κοινότητος. Και αυτό είναι ακεκτημένος δημοκρατίας και πρέπει να το υπερασπιστούμε. Απαντώντας τον κύριο Φαρίας, ο οποίος ανεφέρθη συγκεκριμένα σε αυτό. Εμείς θέλουμε μια ειρηνική και δημοκρατική εξέλιξη επί τη βάση των ελεύθερων εκλογών. επί τη βάση του συντάγματος του 1999, αν ακούσαμε καλά, και εφόσον η εντολή δίδει, που δίδει ο λαός είναι αυτή, πρέπει να ακολουθείτε. Με σεβασμό προς όλους και με απόλυτη συνταγματική νομιμότητα. Ευχαριστώ κύριε Αβελέδο και σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Το θέμα της ε, Βενεζουέλας θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.